λόγος έπειτα από έτοιμα και ηλεκτρονικά και αναλογικά, ε, αναλογικό που θα μπορείτε να, να καταθέσετε στην είσοδο της ε, ε, Ολομέλειας. Κατέφτασε και ο Επίτροπος, οπότε στη θέση του, οπότε του δίνουμε τον λόγο για την εισαγωγική του δήλωση. Mr. President. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων που μου δίδεται η δυνατότητα να σας μιλήσω σήμερα όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι διεξάγεται μία διένεξη η οποία έχει προκαλέσει απέραντη οδύνη για πάρα πολλούς Ισραηλινούς και Παλαιστινίους βλέπουμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται επί τόπου. Έχουμε φαινόμενα βίας, τρομοκρατίας, επέκταση των επικισμών, παράνομη επέκταση των επικισμών και επιπτώσεις ε, της συνεχιζόμενης κατοχής έχουν ε, διαβρώσει την ελπίδα και στις δύο πλευρές και έχουν μειώσει την πιθανότητα βιωσιμότητας μιας λύσης δύο κρατών. Σε διεθνές επίπεδο για πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε καμία ή ελάχιστη ουσιαστικά προσήλωση για την επίλυση της διένεξης αυτής. Και όπως είπε και ένας παρατηρητής πρόσφατα σε μένα πριν από λίγο, δεν υπάρχει ούτε ειρήνη ούτε διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε ενδεχομένω ο μόνο παράγοντας ο οποίο έχει εμπλακεί στην όλη διαδικασία. Με χειρό τρόπο έχουμε υποστηρίξει μια, διαπραγματευ... μια λύση δύο κρατών βάσει διαπραγμάτευση, βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων παραμέτρων και σύμφωνα με το Διεθνές δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι η λύση των δύο κρατών θα πρέπει να βασίζεται στις παραμέτρους εκείνους που βασίζονται σε περάσματα του Συμβουλίου, του δικού μας Συμβουλίου, συμπεράσματα του Ιουλίου του 2014, όπου προβλέπονται οι ανάγκες ασφάλειας του Ισραήλ, καθώς επίσης και η της Παλαιστίνης για ένα κράτος σύμφωνα με τα σύνορα τα οποία προέκυψαν από το 1967. Το δικό μας λοιπόν το όραμα, το ευρωπαϊκό όραμα, είναι ένα όραμα που βασίζεται σε πραγματικές αρχές και είναι και ρεαλιστικό. Αντικατοπτρίζει ουσιαστικά την ευρύτερη προσήλωση που έχουμε ω Ευρωπαίοι σε ένα διεθνές, διεθνή τάξη πραγμάτων που θα βασίζεται σε κανόνες. Επίσης, επεμβαίνουμε επί τόπου. Κανένας άλλος διεθνής παράγοντας δεν έχει εμπλακεί τόσο έμπρακτα προκειμένου να οικοδομηθεί ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα, το 2019 η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της είχαν ένα ανοιχτό ε, ε, ε, είχαν μια χρηματοδότηση, δώσαν 600 εκατομμύρια ευρώ προς τους Παλαιστινίους. Καταλαβαίνετε ότι το ποσό αυτό είναι σχεδόν 1,5 εκατομμύρια την ημέρα χρηματοδοτική βοήθεια προς τους Παλαιστινίους. Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα. Είμαι πεπισμένος ότι ακόμα υπάρχει ένας τρόπος για να σημειώσουμε πρόοδο και για τις δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές θέλουν να ξεκινήσουν αξιόπιστες ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και βέβαια είναι σημαντικό να υπάρχει και διεθνής υποστήριξη για να στεφτεί το όλο εγχείρημα με επιτυχία. Ως προς αυτό λοιπόν, το να υποβάλλονται συγκεκριμένες προτάσεις, όπως το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, θα μπορούσαν να είναι τελικά βοηθητικές προκειμένου τελικά να λειτουργήσουν καταλητικά για να σημειωθεί πρόοδος και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες προκειμένου να ενταθεί η πολιτική ειρηνευτική διαδικασία η οποία έχει αποτελματωθεί εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όπως σας είπα ήδη, η πρόταση που υπευλήθη από τις ΗΠΑ πριν από δύο εβδομάδες ουσιαστικά αντιβαίνει στις διεθνώς αναγνωρισμένες παραμέτρους και είναι πάρα πολύ δύσκολο μέσω της πρότασης αυτής να δει κανείς πώς αυτή η πρωτοβουλία μπορεί τελικά να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εκ νέου. 25 από τα 27 κράτη-μέλη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συμφωνούν με τη στάση αυτή. Δύο χώρες ήταν κατά της άποψης αυτής. Επομένως δεν ήταν η ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου και δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να την παρουσιάσω έτσι. Παρ' όλα αυτά προβαίνω σε μία δήλωση του είπα του εκπροσώπου, την οποία την επαναλαμβάνω και ενώπιόν σα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Ουάσιγκτον και είχα πάρα πολλές ε, επαφές με πάρα πολλούς αξιωματούχους εξωτερικής πολιτικής, υπουργού εξωτερικών, ανώτατους αξιωματούχους επίσης της Αμερικανικής κυβέρνησης. Και έθεσα ακριβώς στους μιλητές μου το ζήτημα αυτό. Του είπα ότι θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Πραγματικά το σχέδιο αυτό αποτελεί βάση για να σημειωθεί πρόοδο ή μήπω όχι. Θα πρέπει ουσιαστικά να γνωρίζουμε αν η πρόταση αυτή καθεαυτή μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, μπορεί να αποτελήσει ένα σημείο κίνησης ή μήπω τελικά αποτελεί ουσιαστικά και το τέλος της όλης διαδικασίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια σαφή θέση. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αναγεννηθεί εκ νέου αυτή η πολιτική διαδικασία προκειμένου να έχουμε μία λύση αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη διεξαγωγή της σημαντικής αυτής συζήτησης, στην οποία είμαι σίγουρο ότι θα συμμετέχετε. Ευχαριστούμε κύριε Μπορέλ. Η συνάδελφος σας έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μπορέλ, είπατε ότι είπα και το σχέδιο τον είπα για τη Μέση Ανατολή από αποτελεί, ε, ε, περιλαμβάνει διεθνείς παραμέτρους. Χρησιμοποιήσατε και μια ιδιαίτερη γλώσσα όσον αφορά το, το ότι αν αυτή η, αυτό το σχέδιο υλοποιηθεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ε, αντιδράσεις. Κάτι που προκάλεσε πράγματι αντίδραση από τους Ισραηλινούς φίλους μας που ε, είπε ότι μπορεί να εξαλειφθεί με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη στάση ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα ε, ο Παλαιστίνιος ε, πρέσβης έχει κατακρίνει το σχέδιο αυτό ως συνωμοσία. Φαίνεται ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν υποδέχεται την πρόταση του Τραμπ με ενθουσιασμό. Όμως εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη και να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Ίσως λοιπόν αυτό το σχέδιο θα μπορούσε να υπηρετήσει ως βάση για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων με ειλικρινή τρόπο και να γίνει κατανοητό ότι θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν επώδυνες υποχωρήσεις. Είναι λοιπόν μια στιγμή που έχετε στη διάθεσή σας κύριε Μπορέλ για να ε, λάμψετε. Η Ευρώπη μπορεί ε, να αναλάβει έναν πιο προβεβλημένο και ειλικρινή ε, ρόλο ως μεσολαβητής και θα μπορούσε να βοηθήσει τις δύο πλευρές να θεωρήσουν αυτό το σχέδιο ως βάση για την έναρξη ουσιοδών διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ασημακοπούλου. Η συνάδελφος Πύρη έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, αγαπητέ εκπρόσωπε της ε, Κομισιόν, δεν ξέρουμε ποιο είναι το όραμα του Προέδρου Τραμπ για τον 21ο ε, αιώνα, εκτός από το ότι είναι παράνομο, μονομερές και προβοκατόρικη προβοκατόρικο. Σίγουρα πάντως δεν είναι μια γνήσια προσπάθεια να εξευρεθεί μια πραγματική και βιώσιμη λύση στην ε, σύγκρουση στην Παλαιστίνη. Οι διαπραγματεύσει μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης σταμάτησαν το 2014. Πρέπει να επαναληφθούν το συντομότερο δυνατόν. Αλλά αυτό δεν είναι ο στόχο του συγκεκριμένου σχεδίου. Ε, το σχέδιο αυτό διαταράσει ε, το διεθνέ σύστημα. Ε, κανόνων. Όχι μόνο νομιμοποιεί τους ε, επικισμούς, αλλά νομιμοποιεί και την παράνομη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης. Πρέπει μια τέτοια προοπτική να γίνει ξεκάθαρο ότι θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις σχέσεις μας με το Ισραήλ. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ανθρώπων. Είτε πρόκειται για ανθρώπους που έχουν χάσει τη γη τους, είτε που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Πρόκειται για ένα κοινικό σχέδιο δύο ακροδεξιών ηγέτες που προσπαθούν να το κάνουν αυτό εν ώψη των εκλογών που έχουν μπροστά τους. Αυτό είναι ένα χαστούκι για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς που θέλουν μια ειλικρινή λύση. Γι' αυτό και σας καλώ, κύριε είπατε εκπρόσωπο, να συνεχίσετε τις προσπάθειες ώστε να εμπλακούν και να, να συμπεριληφθούν όλες οι πλευρές. Οι Παλαιστίνοι και οι Ισραηλινοί χρειάζονται ένα ειρηνευτικό σχέδιο και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαίοι πρέπει να διαδραματίσουμε έναν επικοδομητικό ρόλο στο στόχο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βοτμάντ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι τις περασμένες εβδομάδες και πάλι ε, είδαμε τι θέλει ο κύριος Τραμπ. Λύση δύο κρατών Ισραήλ-Παλαιστίνης με όλα τα πλεονεκτήματα για το Ισραήλ και ψίχουλα για τους Παλαιστινίους. Ένα κράτος θέλει ε, ο Τραμπ και το έχει ε, μεταμφιέσει σε λύση δύο κρατών. Μόνο το Ισραήλ θέλει. Μα είναι εύθραυστη αυτή η σχέση Ισραήλ και Παλαιστίνης. Δεν το αντιμετωπίζει αυτό. Γι' αυτό, κύριε Μπορέλ, θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει. Η, Αμερική τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μονομερή. Έχει τραβήξει το Ισραηλινό χαρτί. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε τη δική μας αξιοπιστία που υπάρχει ακόμα, ενώ η αξιοπιστία των ΗΠΑ έχει κλονιστεί στη Μέση Ανατολή. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ειλικρινείς διαμεσολαβητής, αμερόληπτος. Τώρα θα πρέπει να αρχίσουν οι συνομιλίες Ισραήλ και Παλαιστίνης ξανά. Ε, και αν δεν γίνεται άμεσες, τότε έμεσες διαπραγματεύσεις εκ του συνεγγύς. Είναι απειλή για τη διεθνή κοινότητα αυτό που συμβαίνει. Χρειάζεται μια διεθνής διάσκεψη ειρήνης υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολύ υψηλό επίπεδο. Θα έχετε τη δική μας υποστήριξη προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Βατμάνς. Ένα μισή λεπτό η κυρία Μπον Φρίσκο. Μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, είπατε εκπρόσωπε της Ένωσης, αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ λεπτή και ευαίσθητη η θέση μας. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τη στάση μας, ιδίως γιατί το Βέλγιο, η Εστονία και η Γερμανία ως μη μόνιμα μέλη αυτή τη στιγμή πλαισιώνουν τη Γαλλία και τη στάση της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και με το Brexit τώρα θα πρέπει και εμείς να διεξάγουμε μια εξωτερική πολιτική η οποία να είναι και νέα αλλά και να κοιτάζει όλο και περισσότερο το μέλλον. Να προσαρμόζεται στον 21ο αιώνα που να περνάμε ουσιαστικά περισσότερο από την εξωτερική πολιτική στη μετανάστευση, την ενέργεια, το 5G, την κλιματική αλλαγή αλλά και τις επενδύσεις σε τρίτες χώρες. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει τη δυνατότητα της προώθησης της ειρήνης παντού στον κόσμο. Έτσι λοιπόν όσον αφορά τη Μέση Ανατολή σας καλώ πραγματικά πρωταρχικά να δείτε τρία ζητήματα. Πρώτον, η υπαρξιακή απειλή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Το Ισραήλ είναι ένα εβραϊκό κυρίως κράτος και εμείς οι Ευρωπαίοι στις πιο βαθιές μας αν θέλετε ρίζες είμαστε και εμείς Εβραίοι. Κύριε είπατε εκπρόσωπε λοιπόν, δεν θα πρέπει να χάσετε την καταπληκτική αυτή ευκαιρία να καταδείξετε πραγματικά από ποια πλευρά βρίσκεται η Ευρώπη, σε ποια πλευρά στέκεται η Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Μπομφρίσκο. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο συνάδελφος Beauty Coffer. Πρόεδρε, συνάδελφοι, μεγάλος αριθμός θυμάτων της σύγκρουσης Ισραηλινών Παλαιστινίων ζητούν εδώ και χρόνια ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Ένα τέτοιο ειρηνευτικό σχέδιο βεβαίως και θα πρέπει να περιλαμβάνει επώδυνες παραχωρήσεις και υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές όμως. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ασφάλεια του Ισραήλ, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και ένα βιώσιμο, κυρίαρχο, συνεχές κράτος για τους Παλαιστινίους που ζουν δίπλα-δίπλα με τους Ισραηλινούς. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το σχέδιο του Τραμπ. Δεν είναι μια νέα αρχή, είναι αδιέξοδο. Το αποκαλούμενο σχέδιο ε, ειρήνευση δεν αφορά καν την ειρήνη, γιατί δεν δίνει τέρμα στην σύγκρουση, αντιθέτω την διαιωνίζει. Δεν μπορεί να αποτελέσει βάση διαπραγμάτευσης, αντίθετα αποτελεί ένα σύνολο εντολών. Όταν μιλούν για ειρηνευτικό σχέδιο, στην πραγματικότητα ε, οδηγούν στην προσάρτηση εδαφών άλλο η λύση δύο κρατών και άλλο η λύση ενός κράτους και ενός καντονίου. Ευχαριστούμε κύριε Μπιτικόφα. Ο συνάδελφος Βέμερς έχει το λόγο για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε εκπρόσωπε Μπορέλ καλέσατε και τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και να απόσχουν από μονομερείς δράσεις που θα μπορούσαν να εντείνουν και να οξύνουν ε, την αντιπαράθεση. Αυτή είναι μια στάση η οποία γίνεται αποδεκτή βεβαίως, βεβαίως στο Ισραήλ, αλλά απορρίπτεται από τους Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνοι δεν προσέρχονται καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Πολλοί στον Παλαιστινιακό πληθυσμό προτιμούν τη βία. Στην πραγματικότητα, την ε, τον προηγούμενο μήνα, μη κυβερνητικέ οργανώσει τη Παλαιστίνη αρνήθηκαν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, γιατί υπήρχε ε, κίνδυνο να μην μπορούν αυτά τα χρήματα να καταλήξουν σε τρομοκρατικέ ε, οργανώσει. 75% ε, των μη κυβερνητικών οργανώσεων θεωρούν ότι είναι μπλόφα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε, είπατε εκπρόσωπε, δείξτε σοβαρότητα ω Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεύθυνση της, ε, της ε, ανακούφισης της κατάστασης, της άμβλησης της αντιπαράθεσης και προσπαθήστε να παρακάμψετε αυτήν την στήρα αρνητική στάση που επιδεικνύει η παλαιστινιακή πλευρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Πινέδα για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το δίδυμο Τραμπ ε, Νετανιάχου ε, σε ένα απίστευτο κινησμό ε, παρουσίασαν αυτό το μεγάλο σύμφωνο του αιώνα. Τους Παλαιστίνιους ούτε τους ρώτησαν ούτε υπέγραψαν κανένα τέτοιο σύμφωνο. Παροδία είναι αυτή και παράνομη γιατί παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και άπειρα ψηφίσματα του ΟΗΕ Άρα ούτε συμφωνία είναι, ούτε νόμιμη, ούτε νομιμοποιημένη. Οπότε πόσο μεγάλη συμφωνία του αιώνα. Η μεγάλη απάτη του αιώνα είναι. Και στόχο έχει να ε, εξορροθρεύσει τους Παλαιστινίους και να κρύψει τις ντροπέ δύο εγκληματιών που διώκονται στις χώρες τους. Ο κύριος ε, Μπορέλ πρόσφατα είπε κάτι εξαιρετικό και θέλω να τον ευχαριστήσω. Έχει έρθει η ώρα όμως κύριε Μπορέλ να περάσουμε στα έργα. Φτάνουν τα λόγια. Καλά είναι αυτά που λέτε, αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δράσει και να σταματήσει τη συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ, να αναγνωρίσει το Παλαιπιστηνιακό κράτος, διακόπτει ο Πρόεδρος. Ε, ο κύριος Μάντελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, αξιότιμε Αντιπρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι κάθε δύναμη σε αυτόν τον ε, κόσμο είναι ευπρόσδεκτη αν η δύναμη αυτή εξυπηρετεί την υποβολή προτάσεων για την επίλυση της ε, συγκεκριμένης αντιπαράθεσης, ιδίως όταν πρόκειται για πρόταση με στόχο να επιτευχθεί η λύση των δύο κρατών η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει συμβάλει με συγκεκριμένες προτάσεις σε μεγάλο βαθμό στο παρελθόν. Οπότε νομίζω ότι επικοδομητικά θα πρέπει να προσεγγίσουμε την πρόταση των ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει βεβαίως αναπτυξιακή βοήθεια και άλλα είδη βοήθεια, αλλά δεν έχει προτείνει κάτι συγκεκριμένο στο παρελθόν. Οπότε ας σταθούμε επικοδομητικοί. Αν κάποιο αντιδρά με βία σε μια πρόταση επίλυσης της διαφοράς, τότε αυτός δεν αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και ε, γι' αυτό λέω ότι αυτά θα πρέπει να τα λάβετε υπόψη σας κύριε Επίτροπε, να είμαστε επικοδομητικοί και να είμαστε πάντοτε σε ε, συνεννόηση με τις ε, φιλοδυτικές δυνάμεις αυτού του κόσμου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μάντλ. Για ένα λεπτό ο συνάδελφος Μίξερ. Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε ότι είναι αξιόπιστο το σχέδιο αυτό των ΗΠΑ, καθότι δεν ακολουθεί τι διεθνεί παραμέτρου για την ειρήνη, δεν ακολουθεί τι βασικέ αρχέ του διεθνού δικαίου καν. Και ουσιαστικά μόνο ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνεί με αυτό. Αλλά υπάρχουν, όπω καταλαβαίνετε, και στι ΗΠΑ και στο Ισραήλ εσωτερικοί εθνικοί λόγοι που α, καλούν για την υποβολή ενό τέτοιου σχεδίου που δεν οδηγεί πραγματικά στην ειρήνη οι Παλαιστίνοι έχουν απερίψει το σχέδιο αυτό και ενδεχομένω να ξεκινήσουν βάσει του σχεδίου αυτού τι προσαρτήσει και του επικισμού το Ισραήλ. Τότε στην περίπτωση αυτή θα είναι εντελώ αντιπαραγωγικό το σχέδιο αυτό και ουσιαστικά καταρρύπτει εντελώ οποιοδήποτε ενδεχόμενο λύση δύο κρατών. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει το διεθνέ δίκαιο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προασπίζουμε τη θέση ότι μόνο μία λύση δύο κρατών βάσει διαπραγματεύσεων μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει τι δικαιολογημένε ανησυχίε των Ισραηλινών για ασφάλεια, καθώ επίση και του δικαιολογημένου πόθου για τη δημιουργία ενό κράτου για του Παλαιστινίου. Θα πρέπει επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα αξιόπιστο δικό τη σχέδιο για το πώ θα καταφέρουμε να φτάσουμε τελικά στην πολυπόθετη ειρήνη. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα που φαίνεται τελικά ότι οι ΗΠΑ αποχωρούν όλο και περισσότερο από τη διαδικασία εξέβρεση λύση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Γκέτα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Όταν ο κύριος ε, Τραμπ κάνει λάθος ουσιαστικά με αυτό το σχέδιο ειρήνης, τότε η ειρήνη, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει να κάνει μόνο με το σχετισμό δυνάμεων. Η ειρήνη θα πρέπει να βασίζεται στην ισοτιμία, προκειμένου να έχουμε πραγματικά ένα μέλλον όχι απλώς συνύπαρξης, αλλά συμφιλίωσης. Μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, μόνο υπό την προϋπόθεση αυτή θα υπάρξει πραγματικά μια βιώσιμη ειρήνη. Το βασικό κριτήριο λοιπόν είναι η ισοτιμία και δεν το προτείνετε εσείς αυτό. Δεν πρόκειται λοιπόν να σας ακολουθήσουμε. Θα συνεχίσουμε να λέμε στους φίλους Παλαιστίνους και Ισραηλινούς ότι η Ιερουσαλήμ θα πρέπει να είναι μια κοινή πρωτεύουσα των δύο αυτών λαών που θα πρέπει να έχουν και ασφάλεια και ευημερία. Ορισμένοι θα πούν ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει γιατί έχουμε ήδη κάποια γεγονότα που δεν το επιτρέπουν. Νομίζω όμως θα πρέπει να είμαστε πραγματικά ρεαλιστές. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να κυριαρχήσει είναι η δικαιοσύνη και για τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μάντισον έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ε, Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί τι δύο τελευταίε εβδομάδε ε, είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης, ε, αυτό το σχέδιο ειρήνευση τον είπα για τη Μέση Ανατολή. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να κατανοήσει το, το διεθνές δίκαιο γιατί το διεθνέ δίκαιο προβλέπει το σεβασμό και του Ισραήλ και τη Παλαιστίνης από πλευρά Παλαιστινίων πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν έχουν κατανοήσει ε, το νόημα και την ουσία του διεθνούς δικαίου. Ότι δεν μπορεί δηλαδή να υποστηρίζει κανείς τρομοκρατικές οργανώσεις εναντίον του Ισραήλ. Δεν επιτρέπεται να υποστηρίζει κανείς ε, τον, τον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά σου ως κινούμενες βόμβες για παράδειγμα με βομβιστές αυτοκτονίες εναντίον γειτονικών χωρών. Άρα η Παλαιστίνη παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλοί επικριτέ των ΗΠΑ σχετικά με αυτό το ειρηνευτικό σχέδιο. Αλλά δεν έχω ακούσει και ποτέ καμιά άλλη λύση ή κανένα άλλο σχέδιο ε, για τη Μέση Ανατολή. Οπότε, ο πρόεδρο διακόπτη. Ευχαριστούμε κύριε Μάντισον. Ε, για ένα λεπτό τον λόγο έχει η κυρία Όκεν. Κύριε Μπορέλα, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ρητά είπατε ότι η κατοχή Παλαιστινιακών εδάφων από το Ισραήλ είναι παράνομη. Είπατε επίσης ότι είναι παράνομη και η επικισμοί. Η κατοχή όμως αυτή συνεχίζεται χωρίς να τηρείται καθόλου, να τηρούνται καθόλου τα ψηφίσματα των ΗΠΑ Εθνών. Είπατε ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε τις, την προσάρτηση να συνεχίζεται, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιδράσει, ελπίζω. Το 2016 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα 2334, όπου προβλεπόταν μια δυνατότητα να σταματήσουν οι επικισμοί και να προωθηθεί περισσότερο ο πολιτισμός, οι πολιτιστικές σχέσεις, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν εξελιχθεί εντελώ διαφορετικά. Με τη στάση του το Ισραήλ δεν έχει πραγματικά βοηθήσει καθόλου του Παλαιστινίους, αλλά δεν έχουν αξιοποιηθεί επίση από του Παλαιστινίου τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Δεν επιτρέπω ερώτηση τώρα ενδιάμεση. Προχωρούμε. Ο κύριος Ρέισεν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, αυτή η ειρνευτική συμφωνία έχει απ' όλα. Και φυσικά χωράει και πολύ κριτική. Αλλά ε, σας παρακαλώ σήμερα μην το κάνουμε αυτό. Δεν βοηθάει καθόλου την ενευτική διαδικασία, ούτε την προχωράει κανένα βήμα. Η προστιθέμενη αξία ε, αυτού του σχεδίου είναι ότι βρίσκεται επιτάπητος ε, επιτέλους. Και ας του δώσουμε μια ειλικρινή ευκαιρία. Θέλω να απευθύνω μία και μόνο έκκληση στην Παλαιστινιακή Αρχή. Σταματήστε να υποθάλπετε τρομοκράτες. Αναγνωρίστε το κράτος του Ισραήλ και καθίστε στο τραπέζι να συζητήσετε. Ε, εγώ παίρνω αποστάσεις σαφώς από τα όσα λέει ο ύπατος εκπρόσωπος. Στις 4 Φεβρουαρίου τι κάνατε, μόνο ε, επικρίσεις προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα πρέπει να πείτε στον Αμπάς ότι το καταλαβαίνω ότι δεν θέλετε να διαπραγματευτείτε. Αλλά είναι η λάθος ε, δήλωση, το λάθος μήνυμα. Και γιατί το κάνατε αυτό, εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει ομοφωνία στο Συμβούλιο. Δεν μπορείτε να εκφράζεστε εσείς και να ε, υποτίθετε ότι είναι θέση αυτό της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόισεν. Και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριο Κιζιλίουρεκ. Κύριε Πρόεδρε, η αποκαλούμενη Συμφωνία του αιώνα είναι μια παραβίαση του διεθνούς ε, δικαίου αγνοεί τα νόμιμα συμφέροντα των Πελαισθενείων και προσπαθεί να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα των επικισμών αρνείται τα σύνορα του 67 και αρνείται την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως ε, νόμιμη πρωτεύουσα των Παλαιστινίων. Θα έλεγα ότι το σχέδιο ε, του Τραμπ όχι μόνο παραβιάζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων, η οποία υποσκάπτει το διεθνές δίκαιο συνολικά. Είναι μια επικίνδυνη, απαράδεκτη ε, λύση, πρόταση, όπως αυτή που είχε κατηθεί το 1960. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδείξει αφοσίωση και προσήλωση στην ε, λύση των δύο κρατών στα σύνορα του 1967. Επίσης πρέπει να ε, καταδικάσουμε τους Ισραηλινούς επικισμούς όπως έχουμε κάνει μέσω ε, ψηφισμάτων και να υποστηρίξουμε το δικαίωμα των Παλαιστινίων εκτοπισμένων να επιστρέψουν στις αιστείες τους. Ευχαριστώ κύριε Γιουρέκ. Η συνάδελφος Ινσύρ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ αρνούμαι να χαρακτηρίσω το σχέδιο του Τραμπ ως σχέδιο ειρήνευσης. Πρόκειται για, μια, ε, για ένα σχέδιο ε, πρότασης το οποίο έχει απλώς ε, στόχο να κερδίσει ο Τραμπ τις εκλογές τον Νοέμβριο και να κερδίσει ο φίλος του, ο Νετανιάχου, τις εκλογές στο Ισραήλ αντιβαίνει σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, δεν αναγνωρίζει τα σύνορα του 67, δεν αναγνωρίζει τη λύση δύο κρατών, ε, νομιμοποιεί τους επικισμούς, όλα αυτά σε αντίφαση με την δυνατότητα των Ισραηλινών και Παλαιστινίων να ζήσουν ειρηνικά ως γείτονες. Άρα το ζητούμενο δεν είναι μόνο να μιλάμε εδώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και να αγωνιστούμε για τα δίκαια ε, του Παλαιστινιακού λαού, του Ισραηλινού λαού, να έχει ο καθένας το δικό του κράτος. Εναπόκειται λοιπόν στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναγνωρίσουν επιτέλους την Παλαιστίνη στα σύνορα του 1967. Η Σουηδία το έχει κάνει ήδη, οπότε τώρα θέλω να σας απευθύνω το ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν ώστε να γίνεται σεβαστό το διεθνές δίκαιο από τα κράτη-μέλη της. Ε, ο συνάδελφος Φέστα, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν πήγαινα στο δημοτικό στην Ανατολική Γερμανία, τότε DDR, ε, όπου τότε ε, ήταν υπό σοβιετική διοίκηση προς το παρόν και η Σιλεσία έλεγε προς το παρόν υποπολωνική πολωνική ε, διοίκηση. Αυτό είναι οι χαμένες πατρίδες που νομίζαμε ότι θα ξαναβρούμε. Μόνο ο Βίλι Μπραντ το ε, έληξε αυτό το ψεύμα. Και το ίδιο ισχύει με την ε, Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Ε, αυτοί που ξεκίνησαν τον πόλεμο τον χάσανε και τα πήρε το Ισραήλ. Όποιος ξεκινάει πολέμους αυτά θα πρέπει να τα υπολογίζει. Ε, το μεγάλο ψέμα του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η λύση των δύο κρατών. Η πρόταση του Τραμπ για την ενευτική αυτή προσπάθεια δεν είναι ιδανική, αλλά είμαστε σε αδιέξοδο. Πάνω από 50 χρόνια η Δυτική Όχθη και η Λωρίδα της Γάζας είναι ε, χώροι σύγκρουσης. Εμείς θέλουμε να ε, βαφκαλιζόμαστε ακόμα με τέτοιες χήμερες. Με δύο κράτη δεν υπάρχει λύση. Ευχαριστώ κύριε Φέστ. Ο κύριος Σατούρη. Euh, το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή αποτελεί επικίνδυνη οπισθοδρόμηση, αρνείται το διεθνές δίκαιο, δεν πρόκειται καν για συμφωνία, αλλά ουσιαστικά επαληθεύει μια κεκτημένη πολιτική, πολιτική κεκτημένων μάλλον του Ισραήλ. Εσείς κύριε Μπορέλη πολύ σωστά καταδικάσατε το σχέδιο αυτό. Η κατάσταση όμως είναι πολύ σοβαρή γιατί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν καταφέρνουν ομόφωνα να ζητήσουν την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών χρησιμοποιώντας τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να πετήσουμε από το Ισραήλ να ουσιαστικά αποζημιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση τις καταστροφές που έχει κάνει στα οικοδομήματα εκείνα τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε και εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, διαφοροποίηση ανάμεσα στα αναγνωρισμένα διεθνή σύνορα και τους επικισμούς. Θα πρέπει να καταγγείλουμε και να καταδικάσουμε την επισημοποίηση διακριτικής μεταχείρισης και τέλος και κυρίως πρέπει να πω θα πρέπει να θέσουμε εκ νέου επιτάπητος όπω ζητάνε οι Παλαιστίνοι τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ειρηνευτικής στρατηγικής συνδιάσκεψης για τη Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε κύριε Σατουρή. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η συνάδελφος Φαγιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το σχέδιο ειρήνευσης του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα πραγματικό χαστούκι. Χαστούκι ε, για το διεθνές δίκαιο και για όσους επιδιώκουν να εξευρεθεί μια λύση σε ένα από τα πιο οξυμένα προβλήματα της Μέσης Ανατολής. Δεν υπάρχει περίπτωση να προκύψει λύση μέσα από αυτό το σχέδιο. Πρόκειται απλώ για ένα ακόμη βήμα στην εφαρμογή ενό πλήρου καθεστώτο apartheid, το οποίο το Ισραήλ ήδη έχει επιβάλει εναντίον των Παλαιστινίων. Οι Παλαιστίνοι δεν πρόκειται να αποκτήσουν με αυτό το σχέδιο κυρίαρχο κράτο. Ο Τραμπ προφανώ και δεν συνειδητοποιεί ότι δεν πρόκειται να οδηγηθούμε σε ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ε, ούτε πρόκειται να ε, ε, υπάρξει ειρήνη γενικότερα στην περιοχή αν δεν επιληθεί πρώτα η Ισραηλινο-Παλαιστινιακή διαμάχη και σύγκρουση. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει με ξεκάθαρους όρους να καταδικάσουμε τους επικισμούς, την κατοχή της Δυτικής Όχθης, όλα τα τετελεσμένα των, ε, των ε, παράνομων πράξεων του Ισραήλ. Και θα πρέπει η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τίθεται υπό ε, αίρεση ανάλογα με την συμμόρφωση των Ισραηλινών στα διεθνή πρότυπα. Η κυρία Χουτασάνη. Τα σύνορα του 67 δεν είναι ρεαλιστικά πια, γιατί οι περιστάσεις στην περιοχή έχουν αλλάξει άρδιν τα τελευταία 50 χρόνια. Οι Αμερικανοί είχαν ε, υποσχεθεί να επενδύσουν 50 δις στην, στο ε, κράτος αν εφαρμοστεί το ειρηνευτικό του σχέδιο. Το Ισραήλ επίσης δεσμεύεται ότι δεν θα προχωρήσει σε νέους επικισμούς για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ταυτόχρονα η ε, συνθήκη αυτή, η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει το σχέδιο αυτό. Γιατί ενδέχεται να είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνευσης μετά από πολλές δεκαετίες βίας. Είναι καιρός πια να θέσουμε ένα τέρμα σε αυτή την παρατεταμένη σκληρότατη σύγκρουση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αντιταχθεί σε αυτή την προτινόμενη συμφωνία απλά και μόνο επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μισεί τον Τραμπ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χουκτασάρη. Για ένα λεπτό συνάδελφος ορτάσουν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το σχέδιο του του Τραμπ ε, είναι μονομερές. Ε, βασίζεται στην προσάρτηση, στην αδικία, στην περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και ε, διαιωνίζει την κατοχή και τη σύραξη. Όπως έλεγε προηγουμένως ο συνάδελφος, δεν είναι νευτικό σχέδιο, είναι μια επιταγή. Θέλω να εξάρω το ρόλο του είπα του εκπροσώπου για την ειλικρίνειά του θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική επίλυση μετά από διαπραγμάτευση, λύση δύο κρατών, σεβασμό διεθνού δικαίου και ισότητα των δικαιωμάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρούν την ελπίδα και να την διατηρούν ζωντανή για δύο κράτη και θα πρέπει να αρχίζουν σοβαρά να ε, εξετάζουν το ενδεχόμενο της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους. Θα ήθελα να πω στον είπα το εκπρόσωπο ότι η πολιτική διαφοροποίηση των συνόρων του 67 και τις παράνομες προσαρτήσεις ε, των κατεχομένων θα πρέπει να ε, διατηρηθεί από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση η διάκριση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Ορτάσουν. Για ένα λεπτό, συνάδελφος Μπενιφέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω πολλοί συνάδελφοι, έτσι και εγώ καταδικάζω και αρνούμε το σχέδιο αυτό του Τραμπ για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνη. Πρόκειται για απλή εκλογική προπαγάνδα υπέρ του Νετανιάχου, ο εδώ και μήνε προσπαθεί να κερδίσει μια πλειοψηφία και ουσιαστικά να αποσπάσει την προσοχή των ψηφοφόρων από τι περιπτώσει διαφθορά για τι οποίε κατηγορείται. Το σχέδιο λοιπόν αυτό είναι απαράδεκτο. Καμία διαβούλευση τους Παλαιστινίους δεν άλαβε χώρα. Επίσης βλέπουμε ότι το Ιερουσαλήμ θα είναι αποκλειστική πρωτεύουσα του Ισραήλ, ότι προβλέπεται περισσότερη κατοχή από το Ισραήλ στην Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σωστό το ότι συνολικά απορρίψαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση το σχέδιο αυτό και θα πρέπει να προωθήσουμε τη λύση των δύο κρατών με τα σύνορα του 1967. Σίγουρα οποιαδήποτε μελλοντική προσάρτηση θα έχει πολύ δυσμενεί συνέπειε. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να το πούμε ξεκαθαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποτέ δεν μπορούμε εμεί να σιωπήσουμε μπροστά στην άρνηση της ιστορίας και του διεθνούς δικαίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπενιφέ, Ο συνάδελφος Πίτσουλα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταλαβαίνετε ότι κανένα σχέδιο δεν μπορεί να ευοδοθεί ποτέ και να στεφθεί με επιτυχία αν δεν συμφωνούν και οι δύο εμπλεκόμενε πλευρέ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε απλώ την πολιτική αδυναμία των δύο ηγετών που το προτείνουν. Βλέπουμε την έκφραση μόνο μια μονομερού πολιτική από την κυβέρνηση Τραμπ και τίποτα παραπάνω. Α μην ξεχνάμε πω αντιμετώπισε του Κούρδου, τη Συμφωνία των Παρισίων ή πολλέ άλλε διεθνεί συμφωνίε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ παρουσιάζει ορισμένα ζητήματα ως μια πολύ μεγάλη υποχώρηση από την δική του πλευρά, ενώ ουσιαστικά πρόκειται για μια προσυμφωνημένη πρόταση. Με το Ισραήλ βέβαια μόνο. Επίση, τα όσα λέγονται αυτή τη στιγμή για περαιτέρω προσάρτηση τη κοιλάδα του Ιορδάνη είναι εντελώ απαράδεκτα ή προβλέπεται επίση και η συνέχιση των επικισμών. Όλε αυτέ είναι μονομερεί προσπάθειες και δεν θα οδηγήσουν σε καμία μακροχρόνια βιώσιμη λύση. Η μόνη λύση είναι η λύση των δύο κρατών. Μόνο αυτή η λύση θα επέτρεπε μια ειρηνική συνύπαρξη των δύο αυτών λαών στις δύο πλευρές των συνόρων βάσει πάντα του διεθνού δικαίου. Ευχαριστώ κύριο Σφαίρ στη διαδικασία Κατστιάη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Καλωσορίζω εγώ το σχέδιο, το ειρηνευτικό του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή. Διότι είναι ισόρροπο. Κάτι παίρνουν οι Παλαιστίνοι, την ειρήνη, κάτι ε, παίρνουν επίσης οι Παλαιστίνοι τη χώρα τους και οι Ισραηλοί παίρνουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Οι Παλαιστίνοι απέρριψαν αυτή την προσπάθεια όμως γιατί φαίνεται να τους αρέσει το status quo. Και ρωτώ τώρα τον κύριο Μπορέλ, γιατί ο άλλο που απέρριψε αυτή τη συμφωνία ήταν το Ιράν. Εσείς πρόσφατα είχατε μεταβεί στο Ιράν. Συζητήσατε κύριε Μπορέλ το θέμα αυτό με τους Ιρανούς. Συζητήσατε μήπω και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Και τρίτον, εσείς γιατί πήγατε εκεί. Το μόνο που κάνει αυτό είναι να νομιμοποιεί το καθεστώς που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σφέρ. Ξέχασα να σας πω ότι έχω τριπλάσει αιτήματα για το Catch από τα προβλεπόμενα και παρακαλώ να με συμπαθάτε, δεν θα δώσω σε όλους το λόγο. Ε, κύριος Ρουίθ Ντε Βέσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε είπατε εκπρόσωπε, κύριε Μπορέη. Εγώ στηρίζω το ανακοινωθέν σας και μου φαίνεται σημαντικό και διαδικαστικά για να ξεπεράσουμε τις εμπλοκές στο Συμβούλιο από μία-δύο χώρες. Επί της ουσίας τώρα που είναι το ενευτικό σχέδιο του Προέδρου Τραμπ, δεν θα επαναλάβω αυτό που είπατε εσείς, αλλά και οι περισσότεροι ομιλητέ εδώ για τα προβλήματα που ενέχει, οπότε ε, ότι είναι και αναφάρμοστο. Κάποιοι συνάδελφοι όμως υπενήχθησαν την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή εναλλακτική πρόταση. Αν όχι λεπτομερής πρόταση σαν αυτή που κατέθεσε ο κύριος Τραμπ, ε, ε, ενδεχομένω ε, μια κάποια διαδικαστική πρωτοβουλία, δηλαδή νέα ερευνητική διάσκεψη για τη Μέση Ανατολή, όπως εκείνη που έχει γίνει στη Μαδρίτη το 1991 και αν δεν καθίσταται δυνατό κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, να αρχίσουμε να βάζουμε τα θεμέλια για να υλοποιηθεί στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ροίθ Ντεβέσα. Ο συνάδελφος Στεφανούτσα έχει τον λόγο. Παρακαλώ. Είπατε εκπρόσωπε, κύριε Μπορέλ, εδώ και για δεκαετίες είχαμε διαπραγματεύσει για την ειρήνη και η διεθνής κοινότητα ουσιαστικά προωθούσε μόνο οποιοδήποτε σχέδιο βασιζόταν στο διεθνές δίκαιο αρκεί να ήταν ένα σχέδιο περεκτικό, να βασιζόταν στο διεθνές δίκαιο και να προέβλεπε δύο κράτη για τους δύο αυτούς λαούς που θα μπορούσαν ειρηνικά να συνεπάρχουν και να συμβιώνουν. Καταλαβαίνετε ότι χωρίς ένα τέτοιο σχέδιο δεν μπορούμε να σημειώσουμε πρόοδο. Καταλαβαίνετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί Γι' αυτό συμφωνώ με τον συνάδελφο Βάουτμαν ότι θα πρέπει να έχουμε μια διεθνή συνδιάσκεψη όπου θα εκπροσωπείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια. Νομίζω ότι μια τέτοια λύση πρέπει να προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Στεφανούτσα. Η συνάδελφος Κέμπα έχει το λόγο. Μικρό. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Παρακολούθησα στενά την συζήτηση, αφενός τους ε, υποστηρικτές του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ, αφετέρου τους επικριτές του σχεδίου αυτού δεν υπόθηκαν και πολλά συγκεκριμένα πράγματα σχετικά με το σχέδιο και η δραματική κατάσταση επιτόπου συνεχίζεται. Όποιο ε, έχει βρεθεί στην ε, Ιερουσαλήμ γνωρίζει πόσο δραματική είναι η κατάσταση που επικρατεί, διότι μεγαλώνει μια νέα γενιά η οποία για άλλη μια φορά θα είναι μια χαμένη γενιά. Νομίζω ότι δεν θα ήταν ε, υπερβολή να το πει κανεί αυτό. Οι νέοι άνθρωποι ε, προετοιμάζονται για πόλεμο και όχι για ειρηνική συνύπαρξη. Κύριε Μπορέλ, είπατε ότι έχετε κάνει επαφές με τους εταίρους μας ε, στις ΗΠΑ. Μπορείτε να μας πείτε με ποιον ακριβώς συνομιλήσατε και ποια ήταν τα συμπεράσματα αυτών των συνομιλιών. Γιατί χρειαζόμαστε ένα επικοδομητικό σχέδιο. Είναι αδύρυτη ανάγκη να υπάρξει ένα τέτοιο επικοδομητικό σχέδιο και όποιο θέλει να κάνει επικοδομητικά, επικοδομητικές προτάσεις για σχέδια μπορεί πράγματι να συμβάλλει ώστε να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Η συνάδελφος Μόντικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο ΙΕ έχει διαπιστώσει επανειλημμένος ότι οι επικισμοί αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό το λόγο το σχέδιο των ήπα είναι άκυρο βάσει του διεθνούς δικαίου. Επίσης δεν προβλέπει ε, κυρίαρχο κράτος για τους Παλαιστινίους. Ανεξάρτητα από το σχέδιο το οποίο υποστηρίζει κανείς, δεν μπορεί ένα τέτοιο σχέδιο να αγνοεί το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν δικό τους κράτος. Αντιθέτως, είναι τελείως μονομερές το σχέδιο του Τραμπ που δίνει ε, τα, όλα τα έφορα εδάφη στους Ισραηλινούς και την έρημο στους ε, Παλαιστινίους. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Η πρόταση αυτή είναι ενδεχομένως η χειρότερη που έχει κατατεθεί ποτέ για να επιτευχθεί η ειρήνη στην περιοχή. Ελπίζω ο ύπατος εκπρόσωπος να εργαστεί ώστε ε, και οι δύο πλευρές ε, της σύγκρουσης να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να καταλήξουμε σε μια λύση των δύο κρατών. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Νικολάου Αλαβάνο έχει το λόγο στο τελευταίο στη διαδικασία Κατσδιάη. Δικάζουμε το απαράδεκτο σχέδιο των ΗΠΑ για το Παλαιστινιακό που διαιωνίζει και θωρακίζει την Ισραηλινή κατοχή. Η προωθούμενη συμφωνία εντάσσεται στου υπεριαλιστικού σχεδιασμού των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή. Προβλέπει παραχώρηση τη Ιερουσαλήμ στο Ισραήλ, προσάρτηση τη κοιλάδα του Ιορδάνη και διατήρηση των επικισμών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσει τη και οι ελληνικέ τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάρα πολύ βαριέ ευθύνε κρατούν ίσες αποστάσεις μεταξύ θήτη και θύματος επέκτηναν και αναβαθμίζουν συνεχώς την πολιτική οικονομική στρατιωτική συνεργασία με το ισραηλινό κράτος. η τοποθέτηση του κυρίου μπορέλ που βρίσκει την πρόταση τραμπ συγκεκριμένη και βοηθητική επί της ουσίας έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού ενώ εάν η θέση που εξέφρασε η κυρία Σιμακοπούλου είναι και θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι και απαράδεκτη και επικίνδυνη τέτοιες τοποθετήσεις αποκαλύπτουν τους λόγους που δεν τίθενται σε εφαρμογή οι αποφάσεις κοινοβουλίων που έχουν αναγνωρίσει το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. υποστηρίζουμε το δίκαιο αγώνα του παλαιστινιακού λαού για τερματισμό της ισραηλινής κατοχής για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την ανατολική ιερουσαλήμ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νικόλα Ολαβάνε. Ολοκληρώνεται η διαδικασία Καστιάη. Για να κλείσει ε, τη συζήτηση αυτή θα λάβει και πάλι το λόγο ο κύριος Μπορέλ, υπό τους εκπρόσωπους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους σας. Ξέρουμε ότι αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ διχαστικό και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω ότι εγώ εδώ δεν εκφράζω την προσωπική μου άποψη. Η δουλειά μου είναι να είμαι ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Και χρειάστηκε να εκπροσωπήσω και να εκφράσω αυτό που θεωρώ ότι είναι η γνώμη του Συμβουλίου. Κύριε Σβέρ, δεν είπα εγώ. Δεν είπα εγώ ότι η δήλωση αυτή ήταν θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς είπα, και καλά θα κάνετε να με έχετε ακούσει, ότι ακριβώς επειδή δεν υπήρχε ομοφωνία, το είπα, υπάρχει στα πρακτικά. Εφόσον δεν υπήρχε ομοφωνία, δεν μπορούσα εγώ να παρουσιάσω συμφωνία του Συμβουλίου. Ήταν δήλωση του, είπα, του εκπροσώπου που θα εκπροσωπούσε ποιον. Τα 25 κράτη-μέλη που συμφώνησαν με τη δήλωση αυτή. Το είπα ξεκάθαρα. Εσείς δεν το προσέξατε. Το επαναλαμβάνω. Δεν ήταν δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό. Ήταν μια δήλωση του είπα του εκπροσώπου, διότι δεν υπήρξε ομοφωνία. Κύριε Σβέρ, γιατί πήγα στο Ιράν. Διότι έχω εντολή. Ομόφωνη. Εντολή των κρατών μελών από το Συμβούλιο που μου ζήτησαν να πάω στο Ιράν και να συζητήσω με όλους, γενικά στην περιοχή, την ευρύτερη Μέση Ανατολή, για να προσπαθήσουμε να δούμε αν υπάρχει καμία δυνατότητα για μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεισφέρουμε. Για να αυξηθεί η σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Έχω αυτή την εντολή. Μου είπαν πήγε να μιλήσεις με όλους. Με όλους σημαίνει με όλους. Με τους πάντες. Και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και στην Ιορδανία πήγα και στα Εμμυράτα και στην Τεχεράνη. Θα πάω και στο Ιράκ. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε εκεί να κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι για να βοηθήσουμε, αν μπορούμε στην ειρήνευση και τη σταθερότητα στην περιοχή. Συγγνώμη. Κύριε Σφέρ, δεν με ε, ρωτήσατε εσείς αν ήταν δήλωση ή δήλωση. Έκανα λάθος. Δεν απαντώ σε άλλο συνάδελφο. Ο κύριος Ρόισεν με ρώτησε. Έκανα λάθος. Δεν, ναι, δεν ήταν ερώτηση του κυρίου Σφέρ. Σε εσάς απευθύνεται η απάντηση μου κύριε Ρόισεν. που με ρωτήσατε τι δουλειά είχα στο Ιράν. Φυσικά και μιλούμε με τους Ιρανούς για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και αυτά που απασχολούν ή ανησυχούν και μας. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να διασώσουμε την πυρηνική συμφωνία και τι μπορούμε να κάνουμε για να σταθεροποιήσουμε την περιοχή. Και αφιερώσαμε και πολύ χρόνο στο Ισραηλινό Παλαιστινιακό γιατί βέβαια οι Ιρανοί ξέρουν ότι δεν έχουν και μεγάλο λόγο σε αυτό το θέμα. Η κυρία Κέμπα λέει στι ΗΠΑ με ποιου μιλήσατε. Με τους πιο εξέχοντες. Με τον Υπουργό Εξωτερικών Πομπέο, με του συμβόλους, Εθνική Ασφαλεία, Ασφαλείας, τον κύριο Μπράιαν, με τον κύριο Κούσνερ, τον ίδιο, για το ενευτικό σχέδιο, και με την κυρία Νάνση Πελώση και σίγουρα οι τρεις πρώτοι υποστηρίζουν το δικό του σχέδιο και η κυρία Νάνση Πελώση, όπως γνωρίζετε, ανήκει στους δημοκρατικούς και ήταν πάρα πολύ επικριτική για το σχέδιο αυτό. Όπως σας είπα, εγώ δεν εκφράζω την προσωπική μου άποψη, που είναι και αδιάφορη εν εδώ. Εκφράζω την πλειοψηφία του Συμβουλίου. Και η πλειοψηφία του Συμβουλίου υποστήριξε τη δήλωση αυτή με την οποία στείλαμε ένα μήνυμα λέγοντας ότι πρώτον θα πρέπει οι πάντες να αποφεύγουν τις μονομερείς κινήσεις που στρέφονται κατά του διεθνούς δικαίου και θα μπορούσαν να εντείνουν ακόμα περισσότερο τις κρίσεις και τις εντάσεις και να μην προσαρτηθεί η κοιλάδα του Ιορδάνη. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, μπορεί να είστε βέβαιοι ότι δεν θα είναι ειρηνικό καθόλου. Μπορεί να μην ενδιαφέρει κάποιους, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει πολύ. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε άλλο ένα κέμα βίας στην Παλαιστίνη. Εμείς ζητούμε από τους Παλαιστίνιους να μην κάνουν βίες διαδηλώσεις. Κάναμε μία πρόταση να ξαναδούν τα πράγματα από την αρχή. Αυτό μπορεί να σπάσει το αδιέξοδο και να δημιουργήσει μια δυναμική για να επαναληφθούν και πάλι οι συνομιλίες για το τι μπορούμε εμείς να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Ε, ε, αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ παλιό, πάρα πολύ οδυνηρό και πάρα πολύ επιζήμιο. Δεν αρνούμε να υπάρξει μια νέα αφετηρία. Αυτό που αρνούμε είναι να θεωρείται αυτό τελική έκβαση. Άμα τους πω ελάτε να διαπραγματευτούμε, αλλά θα σας πω ότι αν δεν συμφωνήσουμε θα εφαρμόσω έτσι κι αλλιώς την πρότασή μου, αυτό τι διαπραγμάτευση είναι, ούτε μεγάλο κίνητρο για τη διαπραγμάτευση. Όταν λέμε ελάτε να διαπραγματευτούμε, αλλά αν διαφωνήσετε θα επιβάλλω έτσι κι αλλιώς την πρόταση, αυτό το λέτε εσείς διαπραγμάτευση. Αυτό αρνούμαστε. Και αυτό λέγουμε κιόλα. Και πιστέψτε με, καλέσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών Πομπέων να έρθει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και να εξηγήσει ε, εκ του σύνεγγυς σε όλα τα κράτη-μέλη την πρότασή του. Κάποιοι είναι πιο κοντά σε αυτή την πρόταση, κάποιοι απέχουν πόρο από την πρόταση αυτή και δεν πρόκειται να είναι ομόφωνη η θέση σε αυτό το θέμα. Είναι πάρα πολύ διχαστικό, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε και να κοιτάξουμε να επιδιώξουμε αν όχι την ομοφωνία, τουλάχιστον μια πλειοψηφία που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν το ειρνευτικό αυτό σχέδιο καλή αφετηρία. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θα συνομιλήσουμε με όλους έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να σπάσουμε αυτό το αδιέξοδο και να πιέσουμε για διαπραγματεύσεις. Μερικοί υπεραισιόδοξοι μου είπαν γιατί δεν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι σαν αυτό που έγιναν πολλά χρόνια πριν στη Μαδρίτη, η διαδικασία του Όσλο και της Μαδρίτης. Νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε απλώς να αρνηθούμε λέγοντας ότι δεν είναι καλό αυτό το σχέδιο. Να βρούμε κάτι που να λειτουργεί. Και αυτό θα είναι τμήμα των συζητήσεων που θα έχουμε την άλλη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορέλ. Κλείνει εδώ η συζήτηση αυτή. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ε, δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής και υπά του εκπροσώπου με θέμα την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Συρία. Θυμίζω ότι μπορείτε να ζητήσετε το λόγο με τη διαδικασία της μπλε κάρτας, με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά και τον ηλεκτρονικό. Θα βρείτε σχετικές οδηγίες στην είσοδο της αίθουσας. Αρχίζει και πάλι η συζήτηση με δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής, είπα του εκπροσώπου. Κύριε Μπορέλ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πόλεμος στη Συρία βρίσκεται πλέον στο ένατο του έτος. Πρόκειται για την πιο σοβαρή ανθρωπιστική καταστροφή και κρίση ασφάλειας που ξεδιπλώνεται αυτή τη στιγμή στα βορειοδυτικά της χώρας και σε άλλα τμήματα της Συρίας βλέπουμε αστάθεια και δραματικές ανθρώπινες συνέπειες. Την προηγούμενη Πέμπτη ακούσαμε τον ειδικό απεσταλμένο των ΟΕΕ Εθνών να ενημερώνει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση στο Ιντλίμπ. Περιέγραψαν πως καθεστωτικές δυνάμεις με επικεφαλής το Ιράν και τη Ρωσία έχουν προχωρήσει σε έντονους βομβαρδισμούς χωρίς να ενδιαφέρονται καθόλου για την κατάσταση των αμάχων και για τις υποδομές των αμάχων. Από ό,τι φαίνεται δεν ε, υπάρχει καμία αναλογικότητα. Αυτό είπε ο ειδικό απεσταλμένο των Εθνών. Η ενδυτικοποίηση λοιπόν των στρατιωτικών δράσεων αυτών στο Εντλίπ έχει οδηγήσει σε μια διάκριτη θανάτωση εκατοντάδων πολιτών. Εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι, οι άμαχοι μάλλον να γίνονται στόχοι σε πάρα πολλές περιοχές. Αυτή τη στιγμή ακόμα και καταβλισμοί για τους διεθνούς εκτοπισμένους δέχονται επιθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί μια κατάφορη παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου και θα πρέπει προφανώς οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Οι στρατιωτικέ αυτέ επιχειρήσει ξεκίνησαν στο Εγκλίπ το Φεβρουάριο του 2019, δηλαδή πριν από ένα χρόνο. Και εκ τότε πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί προ την Τουρκία αναφερόμαστε σε ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους ανθρώπους μέσα σε ένα έτος. Και κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι Σύριοι προσπαθούν να διαφύγουν από τις ε, εχθροπραξίες και δεχομένω να έχουμε ένα ακόμα σοβαρό κύμα προσφύγων. Υπάρχουν επίσης αντιπαραθέσεις στρατιωτικές μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και των ε, επισήμων καθεστοτικών ε, συριακών δυνάμεων. Οι εντάσεις αυτές θα μπορούσαν με τη σειρά τους να διευρύνουν ακόμα περισσότερο τη σύγκρουση αυτή στην ευρύτερη περιφέρεια. Η ανακοχή που αποφάσισε η Μόσχα και η Άγκυρα πρέπει να εφαρμοστεί. Έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα, να πω και το ακόλουθο. Μετά από σχεδόν μια δεκαετία βίας, η οδύνη του άμαχου πληθυσμού πρέπει επιτέλου να σταματήσει. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει πλέον τη ζωή του και αυτοί οι οποίοι εξακολουθούν και ζωή αντιμετωπίζουν την προοπτική ενό σκοτεινού μέλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορούμε λοιπόν σε καμία περίπτωση να ανεχθούμε μεγαλύτερη αστάθεια στην περιοχή και μια νέα προσφυγική κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να αποφύγουμε μια αναγέννηση του ΝΤΑΕΣ ή μιας άλλης τρομοκρατικής οργάνωσης στις πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενες αντιμαχόμενες δυνάμεις να εφαρμόσουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και γενικότερα τις παραμέτρους του διεθνούς δικαίου. Ξέρω ότι το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, θα συνεχίζω να το λέω. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι ε, οι πρόσφατες νίκες του Συριακού καθεστώτος δεν μεταφράζονται στα στάθια. Το Συριακό καθεστώς δεν πρόκειται να φέρει ειρήνη και σταθερότητα στη Συρία αν συνεχίσει να ακολουθεί αυτή τη μιλιταριστική στρατιωτική λογική και αν στρέφεται κατά του ίδιου του λαού της. Επίσης, η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο λόγω και της τραπεζικής κρίσης στο Λίβανο. Πρέπει το καθεστώς λοιπόν να αλλάξει πλέον συμπεριφορά αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξ αρχής είχαμε πει ότι μόνο μια περιεκτική σφαιρική πολιτική λύση που ευθυγραμμίζεται με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 22-24 συγκεκριμένα, θα επιτρέψει την σταθερότητα και την ειρήνη στην όλη περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τι προσπάθειε τόσο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών όσο και του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων στα πλαίσια των συνδράσεων τη Γενέβη. Χρειαζόμαστε περαιτέρω επίση ψηφίσματα, καθώ επίση και μία ανακοχή η οποία πραγματικά να υλοποιηθεί στην πράξη. Σας υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και παραμένει ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός δωρητής προς τους Σύριους τόσο εντός της Συρίας όσο και στις κοινότητες των Σύριων προσφύγων στις γειτονικές χώρες. Εμείς υποστηρίζουμε πραγματικά όλους τους άμαχους ε, χαιρετίζουμε την αδεκτικότητά του και θεωρούμε ότι αποτελούν πραγματικά τον κοινωνικό ιστό τη Συρία. Η δική μα λοιπόν υποστήριξη αποτελεί θεμελιώδη επένδυση. Δεν είναι απλώ κάποια χρήματα που δαπανούμε. Είναι ουσιώδη επένδυση στο μέλλον τη Συρία και τη ευρύτερη περιφέρεια, που αποτελεί και μέρο του δικού μα μέλου και ω ε, μέρο του ε, παγκόσμιου συνασπισμού κατά του ΑΝΤΑΕΣ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί τη σταθεροποίηση της κατάστασης στην βόρειο-δυτική Συρία. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα πράγματα, να λάβουμε δράση. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή μέσω του καθεστώτος αυτού να οδηγηθούμε σε μια εξομάλυνση